27 υπέρ και 4 κατά. Συνεπώς εγκρίνεται. Τώρα, οικονομικής 24 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Εκόν 16, οικονομική 16. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οικονομικής 25. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 15-15 απορρίπτεται. Ήτρε 32. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Να επαναλάβουμε γιατί δεν φαίνεται καλά ποιος ψηφίζει υπέρ, ποιος κατά. Ήτρε 32. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας επαναλάβετε για την Ήτρε 32 ψηφίζουμε για να ξέρουμε. Ναι, ναι. Λέω πρόεδρος. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για την τροπολογία 32 της Ήτρε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 11 υπέρ, 20 κατά. Οικονομική 26. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 5. Υπέρ. είπε ο Τρία διορθώνει τώρα. Ήτρε τρία. Υπέρ, κατά, αποχές. Απασχόληση 26. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Απασχόληση 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οικονομική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ΕΚΟΝ 13 θεωρείται εγκεκριμένη. Πάμε στην οικονομική 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίθηκε. Η προηγούμενη. Γιατί κάποιος ρώτησε αν εγκρίθηκε. Τώρα πάμε στην ΕΚΟΝ 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. 27. Ψηφίζουμε για την 27 Ήτρα. Πέρασε ψηφοφορία. 19 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 39 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία Ήτρε 41. Ψηφίστε. 16 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 42 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. της οικονομικής 8 και 9 και της απασχόλησης 24 θεωρούνται εγκεκριμένε. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τώρα συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αναφορών 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αναφορών 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, οι τροπολογίες ε, της οικονομικής 3, 4, 17 και 23 δεν τις ψηφίζουμε διότι έχουν καλυφθεί από άλλες τροπολογίες. Τροπολογία 44 τώρα. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 44. Ψηφίστε παρακαλώ. 17 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. Νομικής, τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ παρακαλώ τους 53. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η οικονομική 10 θεωρείται εγκεκριμένη και τώρα φτάνουμε στη συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αναφορών 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απασχόλησης 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 7 ε, και 9 τώρα τη ΣΥΤΡΕ δεν τις ψηφίζουμε γιατί θεωρούνται εγκεκριμένε. Συμβαστική 11 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 30. Υπέρ, κατά, αποχές, Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για την Ήτρε 30 παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίπτεται. 16-16 είναι το αποτέλεσμα. 63 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 και 65 μαζί τις ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Απασχόληση σε Μα γιατί τις ψηφίζουμε μαζί αυτές τις δύο τροπολογίες. Μπορείτε να μου πείτε. Γιατί εμείς έχουμε διαφορετική ένδειξη. Να ψηφίσουμε διαφορετικά σε αυτές τις δύο. Απασχόληση σε νέα. Υπέρ, κατά, αποχές. Μα πρόεδρε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν απαντήσατε αυτό που σας ρώτησα. Εγώ ρώτησα γιατί τις τροπολογίες 64 και 65 τις ψηφίζουμε μαζί. Γιατί εγώ έχω εδώ ένα κατάλογο ψηφοφορίας που μου δίνει διαφορετική ένδειξη για την κάθε μία. Δηλαδή να ψηφίσω διαφορετικά στη μία και διαφορετικά στην άλλη. Μπορείτε λοιπόν να μου εξηγήσετε γιατί τις ψηφίζαμε μαζί. Εγώ πρότεινα πριν να τις ψηφίσουμε μαζί και ρώτησα αν υπήρχε αντίρρηση. Δεν άκουσα καμιά αντίρρηση. Γι' αυτό. Τώρα βέβαια που ζητάτε το λόγο, παρακαλώ. Μάμα, δεν υπάρχει αντίρρηση τότε να ψηφίσουμε την 65 χωριστά. Αν συμφωνείτε. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Θα κάνουμε το εξή. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 64 και για την 65. Και θα δούμε τότε. Εντάξει. Α, ο κύριος Ταραμπέλα. Όχι, όχι, γιατί εμεί έχουμε ένα πρόβλημα για την 64, ψηφίσουμε διαφορετικά από την 65. Οπότε καλό είναι να ψηφίσουμε χωριστά. Α, αυτό είπατε, α, συγγνώμη, εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ. 64. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 64. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, 65. Υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Απασχόληση σε νέα. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 65. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 3 κατά και 11 αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, απασχόληση 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόληση 10 υπέρ, κα, υπέρ πρώτα, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απασχόληση 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25, τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Της Νομική Επιτροπή 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αναφορών 6 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την ε, αναφορών 6. Λίγη η ψηφοφορία. 19 υπέρ, 13 κατά. Θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Περνάμε στην 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι τραν 1 και έμπλ 17 θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Απασχόλησης 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και η 20 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και περνάμε στην 20, έμπλη 22. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 23. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 67. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ή 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εμπλένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι τραν 10, 11 και 12 θεωρούνται ότι έχουν υιοθετηθεί. Περνάμε στην ε, Γιούρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και περνάμε στη Γιούρι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 69 έχει αποσυρθεί. Έκον 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Απεσύρθη το, η τροπολογία 70, τώρα ψηφίζουμε την 5 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Το 70, η 71 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές. Εβδομήντα πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. η 76 έχει αποσυρθεί και περνάμε στη συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη έμπλ 19 υπέρ κατά αποχές Η 77 απεσύρθη και περνάμε στην Ήτρε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 36. Ξεκινάει η ψηφοφορία, ήτρε 36, λίγη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 13 κατά, έχει εγκριθεί. Η 4 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και περνάμε στην 5. Υπάρχει μία πρόταση, αν συμφωνείτε, να ψηφίσουμε μαζί την ΕΜΠΛ 5, 6, 7, 8 και 25. Εάν συμφωνείτε θα γίνει μία ψηφοφορία για αυτές τις τροπολογίες μαζί υπέρ. Κατά αποχές ενεκρίθησαν. Ε, προτείνω να ψηφίσουμε από κοινού την τραν 2, 4, 5 και 6 σε μία ψηφοφορία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 78 απεσύρθη και περνάμε στην έκον 12 υπέρ, κατά αποχές ενεκρίθη. Έκον 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Για τη 14 ηλεκτρονική, έκον 14, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απερίφθη. Ήτρε 20 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 23 ήτρε υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 25 ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 23, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ήτρε 23, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε λίγοι. 17 υπέρ, 15 κατά, ε, νεκρήθη. είτε 25 θεωρείται ότι έχει οθετηθεί. Περνάμε στην 31 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΙΤΡΕ ε, 26. Ψηφίσατε όλοι, λίγη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 15 κατά, δηλαδή ενεκρίθη. Τραν 9 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Τραν 13 υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. για την τροπολογία ήτρε 38 ο άπαξ και υιοθετήθηκε η Τραν θα ψηφίσουμε μόνο του όρου μέχρι το 2015 υπέρ κατά αποχές απερίφθη η 14 θεωρείται ότι έχει υιοθετηθεί, η 79 απεσύρθη, περνάμε στη συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές. Ενεκρίθη. 80. Λοιπόν, ε, μπορούμε να ψηφίσουμε από την έμπλη 13, 14, 15 και 16 έως 16 μαζί. Όχι. Άρα 13 υπέρ, έμπλη 13 υπέρ, κατά αποχές ενεκρίθη. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 81 για την Ήτρε 11 ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει λίγη 15 υπέρ, 16 κατά, απερίφθη. 81 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη 82 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη έκον 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ ε, ζητήθηκε ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΕΚΟΝ 21 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία έκον 21 ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη. 14 υπέρ 18 κατά απερίφθη. 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Έμπλ αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέχρι το 1 μέχρι 5 οι τροπολογίες της εισηγήτριας μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί υπέρ, κατά. Αποχές ενεκρίθη. Οι τροπολογίες τραν α και β θεωρούνται ότι έχουν υιοθετηθεί και περνάμε στην τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τραν C ε, και D ε, θεωρείται ότι έχει οθετηθεί και περνάμε στην τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ξεκινά. Λίγη. Απερίφθη. 14 υπέρ, 17 κατά. Δεκαπέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε τέσσερα υπέρ κατά αποχές απερίφθηκε. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά. Αποχές. Λοιπόν, έχει υιοθετηθεί η συμβιβαστική 15, θεωρείται ότι έχει Και άρα οι 11, 12, 13, 14 και 16 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθησαν. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για ολόκληρο το σχέδιο του ψηφίσματος. Λίγοι. 32 υπέρ, ε, δηλαδή ομοφωνία. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Θέλω τώρα να ψηφίσουμε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής για το 2013. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρείται ότι ε, εισηγήθηκε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που ηγηθήκατε τη συνεδριάσετος, αλλά σχετικά με την πρόταση αυτή έχω να πω τα εξής. Δεν είναι τόσο προσωπικό, αλλά απευθύνομαι μάλλον στη γραμματεία και βλέπω ότι με τις αλλαγές εις ε, το χρονοδιάγραμμα και στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων ε, υπάρχουν ε, ορισμένες αποστολές που έχουν προβλεφθεί συγχρόνως με τη συνεδρίαση της Επιτροπής εδώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να παραστεί και κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουμε τις πλειοψηφίες οι οποίες εκπροσωπούνται στην Επιτροπή. Εάν λοιπόν λέγεται εγκαίρος μπορούμε ορισμένες ημέρες παραδείγματος 5η 10 ε, Ιανουαρίου που είναι μια εβδομάδα των ε, πολιτικών ομάδων να λεχθεί εγκαίρος ότι δεν θα υπάρχουν ψηφοφορίες αλλά μόνο οι τακτικές συνεδριάσεις της ομάδος. Ε, δεν ξέρω αν δημιουργώ προβλήματα αλλά θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να το επισημάνουμε. Ευχαριστώ. Θα το πούμε στη γραμματεία ώστε να μπορέσει να το κοιτάξει και να κάνει μια καλύτερη διοργάνωση. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι να μην έχουμε συνεδριάσεις πέμπτη απόγευμα. Ε, συμφωνούμε για την πέμπτη το πρωί, αλλά όχι την πέμπτη το απόγευμα. Το σημειώνουμε και θα το φροντίσει η γραμματεία. So let's move, uh, to the... Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο σημείο 10, την έκθεση για την καλύτερη διακυβέρνηση της ενίας αγοράς. Η συγγετής μας είναι ο Ανδρέας Σφάμπ. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο πρώτα στον Ανδρέα και μετά στους σκιώδεις συγγετές. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εδώ μπορώ να αναφερθώ στην ε, ε, έκθεση κατά πρωτοβουλία για την καλύτερη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Πρέπει καταρχήν να σας πω ότι η πρόταση αυτή βασίζεται σε μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε ρητός ότι κατά την εφαρμογή των κανόνων για την ενιαία αγορά ευρύτατα ε, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά εφαρμογής μεταξύ κρατών μελών. Εχθές μιλήσαμε για τον, το ενιαίο ο δίκαιο προστασίας των καταναλωτών με την κυρία Σενάλοβα που εκπροσωπούσε την εισηγήτρια και πρέπει να πούμε ότι πλέον δεν έχουμε ε, δυνατότητα πλέον εφαρμογής και δεν έχουμε πρόσβαση στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς διότι ναι μεν τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο συμβουλίου αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή του δικαίου αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλού υπάρχουν διαφοροποιήσεις και τέλος αλλού δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουμε. Και θα μπορούσα εδώ να αναφερθώ και σε διάφορα παραδείγματα και να αποδείξω ότι στην Ευρώπη και στην ενιαία αγορά έχουμε ένα πρόβλημα στην ενιαία εφαρμογή των κανόνων και των νόμων τους οποίους έχουμε αποφασίσει από κοινού. Ε, πέραν αυτού Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα και εδώ επανέρχομαι διότι εχθές στην ακρόαση σχετικά με το ενιαίο δίκαιο πολίσεων ε, το συζητήσαμε ε, ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν καταστάσεις που είναι συμβιβασμοί με τα κράτη-μέλη και στο τέλος υπάρχει κατακαιρματισμός πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σαν Ευρωπαίοι νομοθέτες δεν έχουμε διαλέξει την καλύτερη δυνατότητα εφαρμογής. Λέω ένα παράδειγμα από τη Γερμανία που έχω συζητήσει με την κυρία Ρούλε. Δηλαδή για το δίκαιο των καταναλωτών στη Γερμανία εφαρμόστηκε το δίκαιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ό,τι ισχύει στη Γερμανία έχει εφαρμοθεί σε μία πρώτη φάση και κάποια άλλη στιγμή Τώρα δηλαδή θα εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία ε, δεν επηρεάζουν θετικά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θεωρούνται ε, σαν ευρωπαϊκή προσαρμογή ενώ το πρώτο μέρος θεωρήθηκε ε, σαν γερμανική προσαρμογή. Δεν υπάρχει ισορροπία λοιπόν ενώ ο Ευρωπαίος νομοθέτης προσπάθησε να καταλήξει σε κάτι αποτελεσματικό και αυτό το λέω διότι δεν ε, ε, θέλω να, να πω ότι βαρύνει περισσότερο η γνώμη του Ευρωπαίου νομοθέτη από τον εθνικό αλλά ότι αν θέλουμε να εφαρμόσουμε την ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι βασικό να υπάρχει ενιαία εφαρμογή και ε, γι' αυτό ο αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να προσέξουμε να γίνεται με τον ίδιο τρόπο η εφαρμογή και γέρος Διαφορετικά βλέπουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας της αυξήσεως κατά 4% της Ευρωπαίας, ευρωπαϊκής αγοράς συνολικά στην επόμενη δεκαετία κατά τρόπον ώστε να φτάσουμε ε, σε ένα ικανοποιητικό ε, επίπεδο. Ε, σύμφωνα με την κυρία Μπάστος της οποίας αποδεχθήκαμε την έκθεση ε, και την ε, έκθεση Γκρέχτ και στην έκθεση της κυρίας Τούν είχαμε συμφωνήσει ότι έχουμε ένα στόχο Δηλαδή ότι οι κανόνες που αναφέρονται στην ενιαία αγορά θα, γίνονται, ε, θα εφαρμόζονται ενιαία. Και γι' αυτό πρέπει να αναλάβουμε ορισμένες πρωτοβουλίες και γι' αυτό σε συζητήσεις με τους συντονιστές συμφωνήσαμε η σημασία της εφαρμογής της ε, του κεκτημένου της ενιαίας αγοράς να είναι τόσο σημαντικό ώστε να καταρτιστεί μία έκθεση κατά πρωτοβουλία και αυτήν σας παρουσιάζω αυτή τη τιμή ε, αυτή τη στιγμή αφού με τιμήσατε και μου την αναθέσατε. Βλέπω λοιπόν και παρουσιάζω τις προτάσεις οι οποίες στο, ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν θα αναφερθούν μόνο στην οικονομική διακυβέρνηση στα κράτη-μέλη αλλά θα χρησιμοποιήσουν ε, και σαν δοκιμασία το, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε. Εξού και σας παρακαλώ ασχέτως των προτάσεων που έχετε κάνει στον τομέα αυτό και που μπορεί να προκύψουν και στο μέλλον να γίνει τώρα μία συζήτηση η οποία κάπου θα καταλήξει γιατί πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ναι έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα τους συγκριτικούς πίνακες παραδείγματος χάρη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή και το, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ε, να προωθήσει μια πιο εύκολη ενία εφαρμογή του δικαίου γιατί αυτό δεν το είχαμε επιτύχει στην πρώτη φάση και είδατε ότι αυτή η διαφάνεια είναι αναγκαία για τους πολίτες και για τη, τα κράτη. Έχουμε προσπαθήσει να υπάρξουν ταχύτερες διαδικασίες α, ε, προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για προφανείς ε, παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου για να μπορέσουν να αποζημιωθούν και, τα ενδεχόμενα, και οι ενδεχόμενες ζημίες και προσπαθούμε να εμπλέξουμε καλύτερα τους ε, Ευρωπαίους πολίτες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για μία σειρά μέτρων την οποία πρέπει να συζητήσουμε από κοινού κατά τρόπον ώστε να ε, ε, οδηγηθούμε σε μία νομοθετική έκθεση και να μην μιλάμε μόνο για την Ευρωζώνη και την μακροοικονομική, τον ε, μακροοικονομικό συντονισμό αλλά οι δημοκρατικές οι δημοκρατικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζονται σωστά και δημοκρατικά και αν αυτό δεν συμβαίνει να δώσουμε μία σαφή ένδειξη στα κράτη-μέλη ε, και ε, να τους εκφράσουμε τη δυσκαρέσκειά μας. Θα επανέλθω για το χρονοδιάγραμμα της εκθέσεώς μου στη συνέχεια αφού ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστούμε θερμά, Ανδρέα. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ την κυρία Μερδάλη, την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς. Θα σας δώσουμε το λόγο αργότερα. Και τώρα θα ακούσουμε τους σκιώδεις συγητές, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ποιος θα κάνει τα σχόλια. Δεν είμαι σκιώδης αλλά θα κάνω πολύ ευχαρίστως κάποια σχόλια. Έγινε μια πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης. Υπάρχει έλλειψη ομοιομορφίας, ομοιογένειας και έλλειμμα στις στην εφαρμογή. Έτσι, χάνουμε 4% ε, δυνητική ανάπτυξη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό δεδομένη της οικονομικής μας κατάστασης. Πρέπει να βελτιώσουμε τις μηχανισμούς εφαρμογής, ε, τη διαδικασία fast track και τη διαφάνεια. Και αυτή μάλιστα τη στιγμή όπου η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το οικονομικό προστατευτισμό κάνει την κατάσταση αυτή ακόμη πιο απαιτητική και επιτακτική ανάγκη να αναλάβουμε κάποια μέτρα. Να υπογραμμίσουμε και τη δέσμευση του Συμβουλίου. Πρέπει να δείξει το Συμβούλιο ότι πραγματικά πιστεύει στην ε, ενιαία αγορά. Γιατί ακούμε τα ίδια τα τελευταία δύο και τρία χρόνια, αλλά έργα δεν βλέπουμε. Πολλά λόγια ακούμε και επένους για την ενιαία αγορά, αλλά δυστυχώς δεν δίνουν την ε, δέουσα σημασία σε αυτή και εμπράκτο στα κράτη-μέλη. Ενώ είναι πολύ σημαντική για την, ελληνική, για την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Χρειάστηκε να δώσουμε μάχη για να ε, αναφέρουμε την σημαντική, τη μεγάλη σημασία και της οικονομίας ε, στα θέματα αυτά για να συμπεριληφθεί και η οικονομία στο εξάμεινο. Δυστυχώς ε, υπάρχουν ελλείψεις στο θέμα αυτό από το Συμβούλιο. Και ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά λένε, αλλά θέλουμε και έργα και κυρίως ε, έμπρακτη αναγνώριση της αξίας με την ε, πρόβλεψη και αντίστοιχων πόρων για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Ο Τόνι Μάντερς απουσιάζει εκ μέρους των Πρασίνων η κυρία Ρούλε. Κυρία Ρούλε, Ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω και να συμπληρώσω σχεδόν όλα που είπε ο κύριος Σφάμπ διότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις οδηγίες αλλά και για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων όπου στο τέλος η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη και πιο δαπανηρή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την τοπική αυτοδιοίκηση Πρέπει λοιπόν ό,τι εφαρμόζεται να είναι εφικτό και για την δημόσια διοίκηση και για τους πολίτες. Και θέλω να υποφεληθώ της ευκαιρίας αυτής να απαιτήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν ε, όσον αφορά την ανάθεση ε, τα delegated η κατεξουσιοδότηση πράξης που έχουμε συμφωνήσει ε, εάν δεν εφαρμόζονται ε, από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το είδα η οδηγία για τις κατασκευές όπου δεν υπάρχει προφανώς έγκαιρη εφαρμογή και παραπονούνται οι ενδιαφερόμενοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πολλές φορές ε, ε, μπορεί να έχει ιδέες για να εξευρωπαίσει την δημόσια διοίκηση των ε, Ευρωπαίων. Πριν δύο χρόνια ήταν το one-stop shop. Το θέμα είναι αν είναι πάντοτε λογικό αν ε, ε, κανείς ε, επιβαρύνει τις ισχύουσες τοπικές διοικήσεις. Τώρα φαίνεται σύγχρονο να υπάρχει μία ανεξάρτητη αρχή για τις δημόσιες προμήθειες και σε άλλους τομείς. Όταν λοιπόν τα κράτη έχουν οικονομική στενότητα και μειώνουν βελτιώνουν τις δομές τους δεν είναι δυνατόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους επιβαρύνει και να τους ζητάει και περισσότερα τέλη. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε και την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ τουλάχιστον έχω διαπιστώσει τουλάχιστον δύο φαινόμενα τα οποία με ανησυχούν. Ευχαριστώ, Ιέμα Μαλ... Μαλ... Μαρκάρκιν από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Η νέα αγορά είναι σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και οικονομική μεγέθυνση. Ε, έχουμε όμω ακόμη πολλού φραγμού στην εσωτερική αγορά και έτσι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το πλήρω δυναμικό τη. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το θέμα τη οικονομική διακυβέρνηση και θα πρέπει να ενισχύσουμε την εφαρμογή, να βελτιώσουμε την εφαρμογή των ε, υπαρχόντων ε, κανονισμών και των υπαρχόντων διατάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύει τα υπάρχοντα εργαλεία και τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Θα πρέπει να τα καταστήσουμε πιο αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και μας ενδιαφέρει μια αιτήσια έκθεση επίδοσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να δούμε πού υπάρχουν τα κενά που χωλαίνει η εφαρμογή και να μην εντοπίσουμε μόνο ε, τα προβλήματα, αλλά να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουν την εφαρμογή. Και φυσικά να μην υπάρχει επικάλυψη μεταξύ του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, αλλά συνεργασία, αξιοποίηση βέλτιστων των πρακτικών και μια σωστή δικτύωση, ώστε να εφαρμόσουμε τις προτεραιότητες της εσωτερικής αγοράς. Και η έξυπνη ε, ρύθμιση είναι προτεραιότητα και φυσικά να προβλέψουμε ε, ειδική μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να επιτρέψουμε εξαιρέσει μόνο αν υπάρχουν αποχρόνοντε λόγοι υπέρ τη ανάπτυξη. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ένα μειόμορφο τρόπο για την κατάθεση παραπώνων εκ μέρου των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταστήσουμε λειτουργική την εσωτερική αγορά. Γιατί όχι και την τεχνολογία, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας για να βελτιώσουμε το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουμε εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Μια ενισχυμένη διακυβέρνηση θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε και την έκθεση για την ενιαία διακυβέρνηση και προσβλέπω σε στενή συνεργασία και με τον εισηγητή και με τους υπόλοιπους και ο εισηγητές γιατί το θέμα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ΚΟΕ, ο Κορνέλης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Ανδρέα Σφάμπ για τις ιδέες που παραθέτει στην έκθεσή του. Το θέμα της διακυβέρνησης εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς, είναι πολύ σημαντικό. Δεν περνάει ούτε μια εβδομάδα που να μην λαμβάνω παράπονα από επιχειρήσει για την έλλειψη εφαρμογή των κανόνων που ήδη έχουμε εγκρίνει. Και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε καλύτερη εφαρμογή, θα συνάδει και στην ε, μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και να επικεντρωθούμε στην υπάρχουσα νομοθεσία. Συμφωνώ. Όταν όμως ε, ε, αναλύω τα παράπονα που φτάνουν σε μένα για την εφαρμογή, διαπιστώνω ότι ίσως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αναλύοντας καλύτερα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανακοίνωση για τα κέντρα της εσωτερικής αγοράς, αλλά να δούμε και το, τους διάφορους μηχανισμούς που έχουμε, Solvit και διάφορους μηχανισμούς ε, επίλυσης των διαφορών Έχουμε πολλές φορές, ε, βλέπω πολλές φορές τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα έχω χαμένα. Πώς να προσανατολιστεί μια μικρομεσαία επιχείρηση. Πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε και την πρόσβαση στους υπάρχοντες μηχανισμούς, να τους απλουστεύσουμε, να τους καταστήσουμε πιο εύχριστους και φυσικά χρειαζόμαστε και έναν ορισμό του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το ρόλο των κρατών μελών σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει μεσολαβητικό ρόλο, αλλά δεν είναι σαφή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ρόλου και των ευθυνών της ε, Επιτροπής αφενός και των κρατών μελών αφετέρου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν ε, απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη με τα οποία έχουμε προβλήματα, ίσω θα πρέπει να το δούμε μέσω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα έχει αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο. Νομίζω ότι και εκεί μπορούμε να βρούμε κάποιε εύχριστε και πρακτικέ λύσει. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπρόσωπο της ε, Ευρώπης για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία, η ΕΦΔ. Άλλος κανείς που θέλει το λόγο. Η κυρία Τάιλερ. Um, uh, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές και τον εισηγητή. Δεν σκόπευα να πάρω το λόγο, αλλά τελικά πιστεύω ότι είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα που θέλω και εγώ να τονίσω κάποια πράγματα που είπαν και άλλοι. Πρώτα απ' όλα το θέμα της επικάλυψης. Αυτό που με απασχολεί είναι η πόροι. Είμαστε σε περίοδο λιτότητας, οπότε η ενιαία αγορά και η νομοθεσία της έχει πολύ σημασία πώς εφαρμόζεται εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ενημερωνόμαστε ώστε να βλέπουμε ποιες χώρες μέλη εφαρμόζουν και ποιες δεν εφαρμόζουν τους κανόνες. Και είναι ενδιαφέρον, τώρα που μιλάμε και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον προπολογισμό, να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η εσωτερική αγορά. Εντάξει, εμεί δεν συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις τις δημοσιονομικές αλλά όπω είπαν και άλλοι ομιλητέ εδώ, η ενιαία αγορά πρέπει να λειτουργεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, αποδοτικά και μόνο τότε μπορούμε να έχουμε και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη την οποία, στην οποία προσβλέπουμε. Τελικά το θέμα είναι οι πόροι. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε εδώ, και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση, το θέμα σας δηλαδή. Οπότε, εν κατακλείδη, το έργο σας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να γίνει σωστά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ότι υπάρχει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και όταν η Επιτροπή λέει ότι οι πόροι δεν δαπανώνται όπως πρέπει στις χώρες μέλη, μα τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 20 χρόνια μετά την ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, προφανώς και θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να δείξουμε ότι τα επόμενα 20 χρόνια θα λειτουργεί η εσωτερική αγορά έτσι ακριβώς όπως τη θέλαμε. Άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Τότε να πω και εγώ τη γνώμη μου. Βλέπω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική πιο σημαντική από ό,τι φαντάζεται κανείς έτσι, όταν την πρωτοδεί. Και αυτό γιατί υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και το ζήτημα της ανάπτυξης. Αν λοιπόν δεν λειτουργεί καλά η ενιαία αγορά, δεν μπορούμε να πετέχουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, δηλαδή αυτά τα οποία περιμένουν από μας οι πολίτες μας και από την Ευρώπη γενικότερα. Έτσι λοιπόν αυτό θα είναι ένα πολύ καλό πακέτο πιστεύω. Και μπορούμε έτσι να συμμετάσχουμε στη συζήτηση για την ε, συμμετοχή της εσωτερικής αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα πρέπει να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια. Και αν θέλουμε να πάμε λίγο πιο μακριά ακόμα, το λέω για να το σκεφτείτε, πρέπει να δούμε πόσο θέλουμε να πιέσουμε τα όρια με τους πίνακες συσχετισμού ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή και εμείς να κάνουμε μια χειρονομία προς τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να πάρουν στα σοβαρά την ε, ομοιομορφία και την ε, εφαρμογή που δυστυχώς βρίσκονται πολύ πίσω ακόμα. Ίσως αυτό να μπορούσε να είναι ένα θέμα μιας μεγάλης συζήτησης ή μιας μελέτης. Πώς το ευρωπαϊκό εξάμεινο δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά στα κράτη-μέλη. Και να το δούμε αυτό και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μερντάλη από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή σας που μου δίνει το λόγο. Ήρθα για να σας μιλήσω για την ανακοίνωση για τη διακυβέρνηση που ετοιμάσαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήρθα επίσης εδώ για να σας πω ότι ειλικρινά με καθισχάσουν πάρα πολύ οι παρεμβάσεις σας, γιατί έτσι βλέπω πόσο σημαντικό είναι το δικό σας έργο, πόσο δηλαδή το δικό σας έργο εδώ στην ΕΜΚΟ μπορεί να βοηθήσει εμάς στην δικιά μας γενική διεύθυνση. Όντως είμαστε σε μια οικονομική κρίση, πάρα πολύ σημαντικό είναι η ανάπτυξη και η ενιαία αγορά αποτελεί τη λύση για την ανάπτυξη. 2.500 νομοθετήματα έχουν να κάνουν με την ενιαία αγορά, καλύπτουν 20 διαφορετικού τομεί ε, σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα. Καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. Εμεί είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια καινοτομία σε έξι διαφορετικού τομεί. Αυτό ακριβώ προτείνουμε εμεί με τη δικιά μα την ανακοίνωση. Και η πρώτη είναι ότι πιστεύουμε πως ορισμένες χώρες μέλη Πρέπει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση για να δουν ολόκληρο το θέμα της ενιαίας αγοράς. Ορισμένες χώρες θα καταφέρουν υπέροχα. Αλλά όταν λέμε μια, ένα κέντρο διακυβέρνησης για την ενιαία αγορά στα κράτη-μέλη, δεν εννοώ μια μαζική οργάνωση τεράστια με δεν ξέρω πόσες θέσεις απασχόλησης. Όχι, λέω, αυτοί που δουλεύουν για την ενιαία αγορά στις χώρες μέλη να συνδέονται μεταξύ τους. Είναι θέμα δικτύωσης δηλαδή, είναι θέμα γνώσης, ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι οι άνθρωποι ε, έρχονται σε εμά και δεν έχουν μεταξύ τους δικτύωση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει κάποιο είδου ε, clearing house, κάποιο είδος δικτύου πας περιπτώσει στις χώρες μέλη για το θέμα αυτό. Τώρα υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Το IMI αρχίζει κάπως κάτι να κάνει που είναι το σύστημα πληροφόρησης για την ενιαία αγορά και καλύπτει όλο και περισσότερα κομμάτια της δουλειάς μας. Ενιαία σημεία επαφής επίσης. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με την πληροφόρηση και τη διαφάνεια. Αλλά είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Άκουσα αυτά που είπατε εσείς για τους πίνακες συσχετισμού. Κανένας ε, δεν ε, λυπάται περισσότερο από εμά για το ότι δεν προχωρήσαμε περισσότερο. Αν είχαμε περισσότερη διαφάνεια και αν έχουμε περισσότερη διαφάνεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μεμονωμένα συστήματα στην Ευρώπη και έτσι να δούμε κατά πόσο γίνεται σωστή εφαρμογή. Οπότε θέλουμε να υπάρξει σύνδεση με τα εθνικά συστήματα και ότι στα εθνικά συστήματα βλέπουμε ποια εθνική νομοθεσία έχει να κάνει με την ενιαγορά. αγορά. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει. Ο τέταρτος τομέας καινοτομίας έχει να κάνει με την επίλυση προβλημάτων. Το solve πρέπει να γίνει καλύτερο, μεγαλύτερο, ευρύτερο και πιο αποτελεσματικό. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και άλλα προβλήματα που τίθενται από πλευράς καταναλωτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εσωτερικών υποθέσεων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Όλοι προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι από την αρχή που ίσως όμως κάποιος άλλος το έχει ήδη επιλύσει. Έπειτα έχουμε το θέμα της, ε, ε, θέσει σε ισχύ, τις εφαρμογές στην πράξη. Λέμε στην ανακοίνωσή μας ότι υπάρχουν 40 διαφορετικές οδηγίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και που είναι κλειδί, υπηρεσίε, ε, προσόντα, ε, συστήματα δικτύωσης, η ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο κλπ. κλπ, κλπ. Είναι κλειδί για την ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι ότι θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να τα αναφέρουμε όλα αυτά, να τα εντοπίζουμε και θα είμαστε και δρακόντιοι όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση μας ε, απέναντι στα κράτη-μέλη. Άμα δηλαδή δεν εφαρμόζεται καλά ε, οι κοινοτικέ ρυθμίσει δεν εφαρμόζονται, θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Πρέπει επίση βέβαια να κοιτάξουμε και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πούμε δηλαδή μήπως τελικά δεν βοηθάμε αρκετά τα κράτη-μέλη όταν ε, τίθεται θέμα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, γιατί και εμείς δαπανάμε πάρα πολύ ενέργεια όπως και εσείς, στη διαπραγμάτευση των ε, νομοθετικών ρυθμίσεων. Μετά, μετά παίρνουμε βαθιά ανάσα και επαναπαυόμαστε. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα όταν φτάνουμε στο στάδιο της ε, συμπερίληψης στην εθνική νομοθεσία του κοινοτικού δικαίου. Και άμα δεν το κάνουμε, εσείς να μας το λέτε. Για να μας μαλώνετε γι' αυτό. Τέλος, θα έχουμε και μία έκθεση για την ενιαία αγορά, η οποία θα συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα επικεντρωθούμε εκεί σε κάθε χώρα μέλος όπου υπάρχουν ελλείψεις. Γιατί βέβαια οι ελλείψεις και δυναμίες είναι διαφορετικές από κράτος σε κράτος. Μπορεί σε μια χώρα κάτι να εφαρμόσετε πάρα πολύ καλά και σε κάποια άλλη όχι. Συνεπώς αυτό για μας θα είναι σημαντικό. Τώρα η μεγάλη δοκιμή θα έρθει όταν θα διαπιστώσουμε κατά πόσο το ευρωπαϊκό εξάμεινο λαμβάνει υπόψη το αυτά που κάνουμε εμείς. Θα δούμε πόσο μεγάλη θα είναι η έκθεση αυτή, πόσα πράγματα θα συμπεριλαμβάνει και πόσο καινοτόμα θα είναι. Και πόσο θα συνδέεται με όλα τα διαφορετικά θέματα, τα έξι τα οποία σας ε, αναφερά που βρίσκονται στην έκθεση για τη διακυβέρνηση θα είναι μια online έκθεση που θα σας δίνει όλες τις λεπτομέρειες. Ελπίζω, αλλά βέβαια εσείς θα το δείτε, ελπίζω κάποια στιγμή να θεσμοθετηθεί ότι μια φορά το χρόνο με τι άλλο θα το κοιτάτε αυτό, θα εντοπίζετε πού είναι τα προβλήματα, πού υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές και να τα συζητάμε αυτά μαζί. Γιατί πραγματικά είναι στοιχεία τα οποία θα είναι πολύ βασικά για να προχωρήσουμε. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Επανέρχομαι τώρα στον Ανδρέα Σφάπ για τα τελευταία του σχόλια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για τα θετικά σας σχόλια όπως και όλα των συναδέλφων που ακολούθησαν το ίδιο σκεπτικό και με τα οποία συμφωνώ ο πλήρως αλλά θέλω σε ορισμένα σημεία να προσθέσω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν με την έκθεση αυτή δεν θέλουμε να δώσουμε ε, την ε, εντύπωση ότι η έκθεση αυτή ανήκει και πρέπει να αναλυφθεί από την ε, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Μπορεί να ε, συμπεριληφθεί και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και άλλες. Ε, επίσης ο Λουίς Κρέχτ μίλησε για uniformity, για ενοποίηση. Εμείς δεν θέλουμε όλα να ενοποιηθούν, αλλά θα θέλαμε στους τομείς στους οποίους στην Ευρώπη θέλουμε να έχουμε μία δημοκρατική νομοθεσία και να έχουμε συνεννοηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με τις κυβερνήσεις ότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν ισότιμα να το διακηρύττουμε και όσον αφορά την επικουρικότητα όταν έχει νόημα πρέπει επίσης ε, να ισχύει σε όλη την Ευρώπη αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο διότι πάντοτε υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα και εδώ δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο αλλά μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις για όλους στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει όλα να ενοποιηθούν στην Ευρώπη ο συνάδελφος Μάντερς που λείπει σήμερα πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότεροι κανονισμοί και λιγότερες οδηγίες και συμφωνώ μαζί του αλλά πρέπει να υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν ε, χρειάζεται να ε, εφαρμοστεί όλο με τη μια. Ε, όσον αφορά τα προϊόντα έχουμε την οδηγία ε, κοινοποιήσεως που προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει τα κράτη-μέλη προτού προβεί σε μία ενοποίηση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα προϊόντα ώστε να μπορέσει να υπάρξει μία αντιμετώπιση από όλα τα κράτη τη μελη Αλλά όσον αφορά την οδηγία κοινοποίησης πρέπει να δούμε αν πρέπει να την επεκτείνουμε πλέον των προϊόντων για να υπάρχει ενιαία εφαρμογή. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή που είπε και η κυρία Ρούλε, είπε ότι πρέπει να τονίσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, και να του πούμε ότι αν θέλει να υποκινήσει και να βελτιωθεί η συνεργασία δεν φτάνει να νομοθετεί αλλά θα πρέπει να είναι πιο συνεπής στην πολύ πιο δύσκολη παρακολούθηση της εφαρμογής μέσω των συναδέλφων της γιατί ε, είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει κανείς μία νέα οδηγία από το να παρακολουθήσει αν εφαρμόζεται σωστά η παλιά. Ε, και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι πιο εύκολο να περάσει μια νέα οδηγία αντί να τσαντίζεται και να ε, καυγαδίζει με ένα κράτος μέλος για το, την ανεπαρκή εφαρμογή της προηγούμενης νομοθεσίας ή της προηγούμενης οδηγίας. Άρα ακόμη και για την ανάθεση θα πω στον κύριο Στόιμπερ ότι και αυτός που ζητούσε να μειωθεί η γραφειοκρατία δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν επαρκώς το ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει κάπως να συμμορφωθούν καλύτερα κατά τρόπον ώστε τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο να μπορέσει να, να σκουμποθεί και να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί διασυνοριακά και μόνο αν συμφωνήσει όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να υλοποιηθεί διότι είναι ένα θέμα το οποίο επεμβαίνει στα εσωτερικά εσωτερικά των κρατών και δεν πρέπει να υποκύψουμε σε εσωτερικά παιχνιδάκια διότι ναι μεν ε, στην ενιαία αγορά έχουν πολλά επιτευχθεί κατά τα τελευταία 20 χρόνια αλλά δεν ε, έχουμε πετύχει τους, όλους τους στόχους μας και αυτό δείχνει ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί κανόνες αλλά δεν υπάρχει ε, κανείς στην Ευρώπη που να εφαρμόζει πραγματικά όλους τους κανόνες και αυτό δεν απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο αλλά σε όλους. Δηλαδή σε όλα τα κράτη ε, υπάρχει σύμπραξη στην ε, ανεπαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας. Άκουσα σήμερα εξαιρετικές ιδέες, θα τις συμπεριλάβω όλες, πρέπει να τις ε, δομήσουμε κάπως καλύτερα και να τις προωθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά χαίρομαι πάρα χάρη πολύ ότι όλοι ομόφωνα ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση. Από πλευράς χρονοδιαγράμματος ε, γνωρίζω ε, μόνο ότι θα ήθελα να το δώσω για μετάφραση, να δώσω για μετάφραση την ε, έκθεση στις 8 Οκτωβρίου και να συζητηθεί το αργότερο το Μάρτιο αλλά με τα μεγάλης χαράς θα ήθελα να έχω τις ιδέες σας για να μπορέσω να τις συμπεριλάβω στην έκθεση που θα καταρτήσω. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Το χρονοδιάγραμμα θα αναγγελθεί στη συνέχεια μετά από συνεννόηση με τον εισηγητή μας, τον Ανδρέα Σφαβ. Ολοκληρώσαμε το σημείο 10 της ημέρης της διάταξης και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Θα δώσω το θα δώσω τη σκητάλη της Προεδρίας στο Λουίς Κρέκ, σε άλλο αντιπρόεδρο, γιατί πρέπει να μεταβώ σε άλλη συνεδρίαση. Θέμα μας είναι η πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Παρακαλώ τον συνάδελφο να με αντικαταστήσει την Προεδρία. Mr. Schwab? Mr. Frank Engel. Mr. Um, Schwab, I understand you'll be replacing Mr. Frank Engel. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα τον κύριο Φρανκ Έγκελ. Σας πειράζει να δώσω κατευθείαν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει την παρουσίαση ο κύριος Νότεμπουμ. Θα μας παρουσιάσει την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Νότεμπουμ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κομέρα να αρχίσει την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Yes, good morning. Thank you for the invitation. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την παρουσίαση με τη Ματάρχης ε, ε, στο Τμήμα Δημοσίων Προμηθειών στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Πρόκειται για ένα κοινό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ε, με επικεφαλή στον Επίτροπο Μπαρνιέ και τη Γενική Διεύθυνση της Αγοράς. Θα γίνει μια κοινή παρουσίαση. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα με την διαδοχή των διαφανειών. Λοιπόν, ποιο είναι το οικονομικό πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε μια γενική διαπίστωση όταν ξεκινήσαμε αυτή την ανάλυση της πρότασης ότι η παρούσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών ε, για τις δημόσιες προμήθειες δεν ήταν ικανοποιητική και μάλιστα υπήρχε μια έντονη διαφορά με τον πολύ ανοιχτό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής αγοράς, της ενωσιακής αγοράς. Και μάλιστα 85% ε, της ευρωπαϊκής αγοράς de facto είναι ανοιχτή σε προμηθευτές επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Βέβαια είναι σκληρός ο ανταγωνισμός των δημοσίων προμηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλουμε αγορές στις καλύτερες δυνατές τιμές. Αυτό είναι το θετικό αποτέλεσμα του σκληρού ανταγωνισμού. Έχουμε όμως δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική πρόσβαση των δικών μας επιχειρήσεων στις αγορές των τρίτων χωρών. Και αυτό φάνηκε στι πρόσφατε διαπραγματεύσει που είχαμε για τη Συμφωνία Δημοσίου Συμβάσεων, τη GPA, που ολοκληρώθηκαν στα τέλη τη προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει τεράστια ανισορροπία μεταξύ των δικών μα δεσμεύσεων απέναντι στου εμπορικού εταίρου και των αντίστοιχων δικών του, που έχουν πολύ μικρότερη πρόσβαση, εξασφαλίζουν πολύ μικρότερη πρόσβαση στην αγορά του. Ένα άλλο φαινόμενο είναι οι αναδυόμενε οικονομίε που αναπτύσσουν ραγδαία τι αγορέ του δημοσίων προμηθειών, αλλά φαίνεται ότι ε, κατευθύνονται προς όλο και μεγαλύτερα περιοριστικά μέτρα στις βιομηχανικέ του πολιτικές θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Σε ό,τι αφορά το μέγεθο ε, τη αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι δημόσιε προμήθειε, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε πάνω από 2-3 εκατομμύρια ευρώ. 370 δισεκατομμύρια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή των ε, οδηγιών, δηλαδή 18,5% του συνολικού μεγέθου τη αγορά δημοσίων προμηθειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα εξασφαλίζουμε πρόσβαση των εταίρων μας ε, του GPA, δηλαδή της ε, Συμφωνίας Προμηθειών ε, Συμβάσεων δημοσίων, δημοσίων Προμηθεών και φυσικά από τους βασικούς μας προμηθευτές, εταίρους μας, συγγνώμη, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες από GPA στην, στο επίπεδο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και 37 πολιτείες και περιορισμένη πρόσβαση σε χαμηλότερα επίπεδα διακυβέρνηση, σε περιορισμένο αριθμό ε, πόλεων με τομεακές Σε Ό,τι αφορά την Ιαπωνία, και εκεί διαπιστώνουμε περιορισμό του πεδίου εφαρμογή ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε. Ε, περιορίζεται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και κάποια επίπεδα υψηλή διακυβέρνηση. Σε χαμηλά επίπεδα διακυβέρνηση ε, που εκπροσωπούν και 500.000 πολίτες δεν συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής. Επίση, με, την υπερβολική χρήση των λειτουργικών ρητρών διασφάλιση, η Ιαπωνία de facto αποκλεί σημαντικού τομεί όπω το σιδηροδρομικό. στον Καναδά, περιορισμένη πρόσβαση σε, σε υπηρεσίες της, δημο, της και, κεντρικής αμοσπονδιακής κυβέρνησης. Έχει περιοριστεί και η πρόσβαση σε, κεντρικά, ε, σε κεντρικούς ε, οργανισμούς, ε, αλλά κάποιων πόλεων, αλλά όχι σε κοινοφελείς επιχειρήσεις όπως είναι οι σιδηρόδρομοι και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες. Στην Κορέα επίσης υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε αγαθά που καλύπτονται από την GPA. Ε, αποκλεί η Κορέα 75 πόλεις, 86 κομιτείες και 69 αυτόνομες περιφέρειες. Τέλος έχουμε την Κίνα που αυτή τη στιγμή μια και δεν ούτε στην GPA ούτε σε οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, de facto ολόκληρη της αγορά είναι κλειστή. Και μάλιστα 83 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2007 και έκτοτε έχει εξελιχθεί ραγδαία φυσικά. Έχουμε πολλούς περιορισμούς που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Υπάρχει νομοθεσία που δίνει σημαντική προτεραιότητα στα τοπικά προϊόντα. Επίσης υπάρχουν ε, υποχρεώσεις τοπικού περιεχομένου μέχρι 50% και αν δεν τηρηθούν αυτές εφαρμόζονται περιορισμοί στις τιμές ή προτιμησιακές τιμές και επίσης προβλέπουν την ad hoc δυνατότητα στο δίκαιο δημοσίων προμηθειών να αυξήσουν την υποχρέωση για τοπικό περιεχόμενο μέχρι και 70%. Οπότε, αν συγκρίνουμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις των πέντε σημαντικότερων εμπορικών εταίρων, καταλήγουμε σε αυτά τα στοιχεία που εξασφαλίζουν ε, την εγγυημένη πρόσβαση στην αγορά και δεν λαμβάνει υπόψη την de facto κατάσταση που για την Ευρώπη είναι πολύ πιο δυσμενής και καλύπτει ε, για την Ευρώπη περίπου 95% πρόσβαση στους εξοκοινωτικούς εταίρους, κάτι που δεν ισχύει. Το αντίστοιχο δεν ισχύει από την πλευρά των εμπορικών εταίρων. Βλέπετε επίσης ε, τη σύγκριση των 12 βασικών μας ε, ε, εταιρών, 25% ε, καλύπτεται μέσω του GPA και άλλων ε, FTA. Υπάρχει το εγχώριο άνοιγμα, η de facto κατάσταση δηλαδή, παρόλο που δεν υπάρχει συμφωνία, επιτρέπουν πρόσβαση στην αγορά σε άλλο αλλοδαπές εταιρείε. Το τρίτο τμήμα είναι η παράκαμψη των τοπικών εμπορικών φραγμών για φαρμακευτικά προϊόντα, για παράδειγμα η κάποιο εξοπλισμό για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, για τα αεροδρόμια. Πολύ συχνά εκεί οι επιχειρήσει παρακάμπτουν το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγγυημένη δέσμευση εξαιτία της υψηλής εξειδίκευσης που απαιτείται για τα προϊόντα αυτά, αλλά παρόλα αυτά 53% της αγοράς δημοσίων προμηθειών μπλοκάρεται ε, μέσω των τοπικών εμπορικών φραγμών. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό και νομικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο δύο ε, νομοθετικά τμήματα που αναφέρονται σε τρίτες χώρες. Το άρθρο 58 της Οδηγίας για τις Κοινοφελείς Υπηρεσίες που προβλέπει ότι οι αναθέτοντες φορείς μπορεί να απορρίψουν προσφορές που περιλαμβάνουν πάνω από 50% αλλοδαπών προϊόντων και το, η σκέψη 18 ε, που προβλέπει δυνατότητα αποκλεισμού τρίτων χωρών για προμήθειες που δεν αφορούν την άμυνα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ε, μια νομική πρόταση, δεν ε, προβλέπει νομικές διατάξεις σε ό,τι φορά την μετάθεση στην κοινωτική νομοθεσία των ε, περιορισμών ή των επιφυλάξεων που έχουμε διαπραγματευτεί με τους εταίρους. Οπότε, οπότε, χάνουμε δυστυχώς ε, πολλές ε, εξαγωγές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπολογίζονται σε 4 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης έχουμε περιορισμένη δυνατότητα των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος, σε αντίθεση με τους εμπορικούς μας εταίρους που έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στις δικές μας αγορές. Οπότε οι εμπορικοί μας εταίροι μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος, να ε, ομαδοποιήσουν τις επενδύσεις και να προσφέρουν πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές στις τρίτες αγορές. Επίσης, λαμβάνονται στρεβλωμένες επιχειρησιακές αποφάσεις. Γιατί σε ορισμένες χώρες η πρόσβαση de facto εμποδίζεται. Γιατί υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να έχουν ε, τοπική έδρα όταν ε, ε, ασχολούνται με μεταφορά τεχνογνωσίας. Οπότε θα πρέπει τα οι νομοθέτες να τους πούν αν πραγματικά έχει νόημα μια τέτοια απόφαση επιχειρηματική δημιουργείται μια de facto κατάσταση αθέμητου ανταγωνισμού, έλλειψη ηθικών ίσου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με τι επιχειρήσει των βασικών μας εμπορικών εταίρων. Ποιοι είναι οι στόχοι μας λοιπόν. Αυτή είναι η στόχη που προσπαθήσαμε να ελοπίσουμε στην, ε, στην προσπάθεια υποβολή μια νέα πρόταση. Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο, ένα μηχανισμό που θα ενισχύει τι εξαγωγέ Ευρωπαϊκή Ένωση τι αγορέ δημοσίων προμηθειών εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε την άσκηση επιρροή Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μόχλευσή τη δηλαδή στι διαπραγματεύσει. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε... των τρίτων χωρών στη δική μα αγορά και να εξασφαλίσουμε την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Μεταξύ των ε, πολιτικών επιλογής που αναλύσαμε ε, είναι η εξή. Καταρχήν έχουμε το βασικό σενάριο. Το σενάριο αφετηρίας, δηλαδή στα τουκβό, συνεχίζουμε με την παρούσα κατάσταση. Όπως λέει και η μελέτη αντικτύπου δεν νομίζω ότι με μια τέτοια επιλογή θα επιλύσουμε κανένα πρόβλημα. Δεύτερη ε, πολιτική θα ήταν μη ε, νομοθετικές, μη δεσμευτικές ε, ρυθμίσεις, δηλαδή soft law, χρήση των άρθρων 58 και 59 της Οδηγίας για τις κοινοφελείς υπηρεσίες, χρήση ταυτόχρονα εσωτερικών και εξωτερικών διεθνών διορθωτικών μέτρων και διεύρυνση των διεθνών διαπραγματεύσεων. Και πάλι όμως για τις επιλογές αυτές το συμπέρασμα ήταν ότι δεν θα ενίσχυαν την επιρροή μας στις διαπραγματεύσεις, ούτε θα βελτίωναν την παρούσα κατάσταση, ούτε θα μας εξασφάλιζαν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές δημοσίων προμηθειών των τρίτων χωρών. Μία τρίτη επιλογή που εξετάσαμε είναι κάποια νομοθετικά μέτρα και έχουμε εδώ διάφορες υποκατηγορίες. Ε, η πρώτη υποκατηγορία, η λύση 3α, είναι να εφαρμόσουμε όλες τις, ε, τους περιορισμούς ε, που διαπραγματευθήκαμε. Δηλαδή, αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι με τους εμπορικούς μας εταίρους και βλέπουμε ότι εκείνοι είναι απρόθυμοι να ανοίξουν έναν συγκεκριμένο τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει «Α, εσείς δεν ανοίγετε το σιδηροδρομικό σας τομέα, τότε δεν μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε πρόσβαση στο δικό μας σιδηροδρομικό τομέα». Βέβαια το θέμα είναι ε, διαπραγματευτικό, γιατί είχαμε, υπήρχε ίσως ε, νομικό δικαίωμα, αλλά δεν ασκήθηκε αυτό το δικαίωμα. Βέβαια, έτσι ίσως καταλήγαμε στην περίεργη κατάσταση όπου χώρες που δεν έχουν καμία διαπραγμάτευση μαζί μας να έρθουν σε χειρότερη ε, θέση από αυτούς με τις οποίες διαπραγματεύσαμε, διαπραγματευτήκαμε και να έρθουν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Επίσης, ε, στις δημόσιες διαβουλεύσεις είχαμε σαφή διαφωνία μεταξύ δύο πλευρών. Η μία ήθελε πολύ πιο περιοριστική λύση και η άλλη πολύ πιο χαλαρή και πολύ λιγότερο περιοριστική λύση. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε μια χρυσή τομή, μια εναλλακτική που θα μπορούσε να συγκεντρώσει συμφωνία και από τις δύο πλευρές. Και καταλήξαμε στην εναλλακτική λύση 3β. Εδώ έχουμε ε, κάποια βασικά εργαλεία. Πρώτον, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απορρίψουν μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες και όταν λέμε μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες, εννοούμε υπηρεσίες και αγαθά για τις οποίες δεν έχουμε νομικές υποχρεώσεις, δεν καλύπτονται από διεθνείς συμφωνίες. Οπότε δεν έχουμε νομική υποχρέωση σε τρίτες χώρες να τους εξασφαλίσουμε πρόσβαση υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό αποφασίστηκε για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι θέμα εξωτερικής εμπορικής πολιτικής. Οπότε καλό θα ήταν να εξασφαλίσουμε μια επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφύγουμε παρερμηνία των διεθνών μας ε, υποχρεώσεων και να αποφύγουμε φυσικά να αντιμετωπίσουμε νομικά προβλήματα. Γιατί είναι πολύ εύκολο με τις παρερμηνίες να βρεθούμε σε στραβό δρόμο. Επίσης ένα κεντροποιημένο μηχανισμό που προβλέπει μια διαβούλευση, έρευνα και ενδεχομένως επιβολή περιοριστικών μέτρων και πάλι, επαναλαμβάνω, για μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες από διεθνείς συμφωνίες. Μία άλλη επιλογή είναι να επεκτείνουμε την προηγούμενη επιλογή σε αναθέτουσες αρχές ώστε να δέχονται μη καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλους τομείς. Επιλογή 4 παράταση ή παρέκταση των άρθρων 58 και 59 στο πλήρες πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες για να καλύπτουν και τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Επιλογή 5. Επιβολή ενός συστήματος προτίμησης 25% δηλαδή αγοράστε ευρωπαϊκά. Άλλες χώρες έχουν παρόμοιες πολιτικές. Και η επιλογή 6 να, να διορθώσουμε τις ε, άδικες και ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Αυτό το επισημάνουμε στις περσινές μας διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Τώρα σε ό,τι φορά τον αντίκτυπο, την αξιολόγηση αντικτύπου, ως προς τη μεθοδολογία, σκεφτήκαμε ότι από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε. Δεν είχαμε δεδομένα στη διάθεσή μας. Αυτό που έγινε στην αξιολόγηση του αντικτύπου είναι καταμετρήσαμε την ξένη διείσδυση σε κοινοτική αγορά δημοσίων προμηθειών και ταυτόχρονα τη διείσδυση ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αλλοδαπές αγορές δημοσίων προμηθειών. Επίσης είδαμε πόσο μεγάλες ήταν οι αγορές προμηθειών στις διάφορες ε, χώρες και κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσωμείωση αναλύσαμε 22 τομείς προτεραιότητας δημοσίων προμηθειών. Είδαμε ποιες, ποιοι τομείς είναι κλειστοί στις τρίτες χώρες, ποιοι είναι ανοιχτοί, πόσο αξιόπιστη είναι η βιομηχανία στις χώρες αυτές ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Και φυσικά πρέπει να, χρησιμο... να υπολογίσουμε και τη μόχλευση, την ε, επιρροή που μπορούμε να ασκήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Σκεφτήκαμε ότι όσο μπορεί κανείς δυνητικά έστω να μπλοκάρει την αγορά του, τόσο περισσότερο ε, δίνει ενάυσματα στον ε, εμπορικό εταίρο για διαπραγματεύσεις. Οπότε, αν ε, ενδιαφέρονται για την αγορά, για ανατομία τομέα της αγοράς και δεν έχουν εξασφαλισμένη εγγυημένη πρόσβαση, έχουν μεγαλύτερο συμφέρον για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Τρεις παράμετρα χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση των στόχων, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η συνοχή. Και μάλιστα προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αυτές τις τρεις παραμέτρους σε νέα κριτήρια. Ε, Το αντίκτυπο ε, στο εμπόριο και τις, και τις θέσεις απασχόλησης, ανταγωνιστικότητα, μόχλευση, διασάφηση κανόνων, οικονομικά, διοικητικό άγχος, αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και την καινοτομία, στους καταναλωτές, περιβαλλοντικός αντίκτυπος και όταν συγκρίναμε τις διάφορες επιλογές είδαμε ότι η πρώτη επιλογή δεν υλοποιούσε κανέναν από τους στόχους που είχαμε θεσπίσει. Οι επιλογές 2 και 5 πραγματοποιούν κάποιους στόχους, αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και περιορίζουν και έχουν περιορισμένη αύξηση όμως των δυνητικών ε, εξαγωγών οι επιλογές 3α, 3γ και 4 κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιήσουν τους στόχους, αλλά επειδή υπάρχει πιθανότητα για μεγάλο κόστος αντικτύπων, ίσως τελικά δεν είναι πιο αποδοτικές. Η επιλογή 3β είναι η πιο πιθανή να πραγματοποιήσει τους περισσότερους στόχους και έχει και τις καλύτερες επιδόσεις με βάση τις τρεις παραμέτρους μας, ενώ η επιλογή 6 είναι η μόνη που μπορεί να αντιμετωπίσει το, τις ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές και ένα πεδίο ίσου ανταγωνισμού και θεμητού ανταγωνισμού στην αγορά δημοσίων προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περάσω τώρα στην πρόταση που έχουμε καταθέσει και για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, γιατί ένα ξεχωριστό νομικό εργαλείο. Μια και η πρόταση αυτή καλύπτει το θέμα της πρόσβασης στην αγορά δημοσίων ε, προμηθειών της Ευρωπαϊκής Αγοράς από τρίτες χώρες, θεωρήσαμε ότι η κατάλληλη νομική βάση είναι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα έχουμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο και μια νομική βάση για το κείμενο αυτό. Και για να εξασφαλίσουμε ένα ενιαίο πλαίσιο, αποφασίσαμε να προτείνουμε κανονισμό και όχι οδηγία. Ήταν ένα από τα προβλήματα που διαπιστώσαμε ήταν η άνηση εφαρμογή των οδηγιών στον τομέα αυτό από τα διάφορα Πέραν των ορισμών και του συνήθους περιεχομένου, στον κανονισμό αυτό προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε τους κανόνες. Και φυσικά ένα τέτοιο νομικό εργαλείο έχει δίνει ένα σημαντικό μήνυμα προς τις τρίτες χώρες, οπότε από την αρχή θα έπρεπε στο, έπρεπε στο άρθρο 4 να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα καλυπτόμενα αγαθά και υπηρεσίες ε, θα τύχουν ίσης μεταχείρισης με τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν είναι πρόκειτο να κλείσουμε τις αγορές μας, αλλά ότι είμαστε πρόθυμοι να σεβαστούμε όλες τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Ταυτόχρονα έχουμε και το άρθρο 5 που θεσπίζει την αρχή του ανοίγματο. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας ε, ε, ενώ οι εμπορικοί μας εταίροι δεν έχουν ως βασικό σενάριο το άνοιγμα, σε περίπτωση που δεν προβλεφθεί κάτι διαφορετικό, εκτός και αν εφαρμόζονται τα άρθρα 6 ή 8 με 10 που προβλέπουν κάποιους όρους. Και το πρώτο από τα δύο εργαλεία που προτείνουμε είναι το άρθρο 6, το αποκεντρωμένο, εργαλείο που υπάρχει δυνατότητα σε αναθέτουσες αρχές να αποκλείσουν αλλοδαπές προσφορές ε, που δεν καλύπτονται αν υπερβαίνουν το κατόφλι των 5 εκατομμυρίων ευρώ και αν υπάρχει το 50% των μη καλυπτόμενων αγαθών. Φυσικά τον τελικό λόγο για, τις, ε, για τον αποκλεισμό αυτό τον έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερος πυλώνας της πρότασης, το δεύτερο εργαλείο, είναι το κεντρικό, το συγκεντρωτικό εργαλείο που παρατίθεται στα άρθρα 8 με 10. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, ακόμη και όταν ξεκινήσει μια έρευνα. Ποια είναι λοιπόν τα διάφορα βήματα. Με απλά λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε αυτεπαγγέλτος με δική της πρωτοβουλία, είτε με τα αίτηση των κρατών μελών ή από ζήτημα κάποιου ενδιαφερόμενου λάβει την πληροφορία ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης αγοράς στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, τότε μπορεί να ξεκινήσει μια έρευνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διαλευκάνει τους όρους πρόσβασης στη συγκεκριμένη αγορά του τρίτου μέρους. Και μετά την έρευνα γίνονται διαβουλεύσεις με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Τώρα αν αυτές οι έρευνες καταλήξει το συμπέρασμα ότι όντω υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην πρόσβαση της αγοράς, το επόμενο στάδιο είναι να προσκαλέσουμε αυτή την τρίτη χώρα για να διαπραγματευτούμε μια λύση και να βελτιώσουμε την πρόσβαση ε, της αγορά, στην αγορά της. Και εφόσον οι διαπραγματεύσεις αυτές είτε να βαγίσουν είτε απορριφθούν από το τρίτο μέρος, τότε υπάρχει η ε, τη δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει και να θεσπίσει περιοριστικά μέτρα κατά της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, περιορίζοντας τη δική της πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Αγορά ή να επιβάλλει κάποια πρόστιμα χρηματικά αντίπεινα που θα είναι φυσικά ανάλογα με το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί στην αγορά της τρίτης χώρας. υπάρχει και το συμπληρωματικό εργαλείο που περιγράφθηκε στην έκτη επιλογή και είναι το μόνο εργαλείο που μπορεί να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Συνδυάζεται με κάποια άρθρα της αντίστοιχη οδηγία για τις ασυνήθιστες χαμηλές τιμές και όπως έμεσα στο άρθρο 69 θέλουμε να, να κάνουμε τη σωστή διάγνωση κατά πόσο μία προσφορά, η ιδιαίτερα ασυνήθιστη χαμηλή προσφορά, μπορεί να παρέχει να παράσει τα προϊόντα που ισχυρίζεται ότι θα προμηθεύσει με βάση αυτή την ασυνήθιστα χαμηλή τιμή. Σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου δεν διαθέτουμε μια περιεκτική εξωτερική πολιτική δημοσίων προμηθειών και έχουμε και, μια, και ένα κατακαιρματισμό. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις με μονομένα κράτη-μέλη ε, αυτενέργησαν και αυτό δημιουργεί ένα κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς και έτσι μειώνεται και η διαπραγματευτική μας ισχύ στις διαπραγματεύσεις. Μειώνεται η επιρροή μα. Οι εμπορικοί μα εταίροι δεν είναι πρόθυμοι να ανοίξουν τις δικέ του αγορές εφόσον έχουν πληροφορίε για περιορισμού σε αγορές ορισμένων χωρών μελών. Έτσι έχουμε μια κατακαιρματισμένη εσωτερική αγορά και έναν ενισχυμένο κίνδυνο προστατευτισμού. Ορισμένοι εμπορικοί μας εταίροι θέλουν να υιοθετήσουν όλο και περισσότερα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς τους για τις ντόπιε επιχειρήσεις τους. Θέλουμε λοιπόν με την πρόταση αυτή μια πραγματικά περιεκτική και συνολική εξωτερική πολιτική δημοσίων προμηθειών που θα μιλούμε όλοι με ενιαία φωνή, θα αυξήσουμε, θα ενισχύσουμε την άσκηση επιρροής μας στις διαπραγματεύσεις γιατί μερικές φορές ήταν πολύ δύσκολες αυτές για να εξασφαλίσουμε άνοιγμα των αγορών των εμπορικών μας εταίρων και θα εξασφαλίσουμε και ένα θεμητό ανταγωνισμό, ένα fair play, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Ακόμη και ο κλάδος ζήτησε μερικές φορές δραστικά μέτρα. Θέλουμε να δείξουμε όμως ότι δεν είμαστε κατά του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην έρθουν σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση οι δικές μας επιχειρήσεις σε αγορές τρίτων χωρών. Και αυτό ήταν ένα από του στόχου και μια δυναμία που προσπάθησε να καλύψει η πρότασή μα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για την τόσο ξεκάθαρη και τόσο αναλυτική παρουσίασή τους. Και πρέπει να σας πω ότι με εξέπληξε ο τρόπος με τον οποίο οι γενικές διευθύνσεις πέρασαν η μία το λόγο στην άλλη. Τόσο έτσι ήπια, τόσο ωραία. Ο κύριος Βάπ τώρα παρακαλώ να μιλήσει στην Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σήμερα αυτό είναι πολύ θετικό ότι μπορούμε να ε, έχουμε μία πιο εκτενή πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το υπόβαθρο αυτής της πρότασης γιατί όσοι έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα είπαν ότι υπήρχαν διαφορετικά και απόψεις και συνειδητοποιήσεις για το τι μπορεί να επιτύχει αυτή η πρόταση διότι υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στην Ευρώπη. Από τη μία πλευρά λέγεται ότι διεθνώς κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να απορρίψουμε την, ε, ε, την ευπιστία μας και να ισχύσει η Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Απλούστατα δίνουμε προστατευτικά μηνύματα ε, και αποκαρδιώνουμε τους ομολόγους μας στον εμπορικό τομέα. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή την Επιτροπή πρέπει να φροντίσουμε στο το θέμα αυτό, να τονίσουμε περισσότερο τα στοιχεία τα οποία προωθούν την ε, ε, ενιαία αγορά και που δεν προωθούν την γραφειοκρατία και γι' αυτό θα αναφερθώ στο άρθρο 6 το οποίο μόλις παρουσιάστηκε το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις ε, ε, αρχές οι οποίες ε, αποφασίζουν για τις δημόσιες προμήθειες να αποκλείσουν από τις διαδικασίες της εταιρείε των χωρών που δεν έχουν υπογράψει το GPA και όπου η προσφορά περιέχει στοιχεία εκ των οποίων τουλάχιστον το 50% δεν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όντως μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει τα βλέπουμε όλα αυτά αλλά εγώ αναρωτιέμαι πώς θα μπορεί η αρχή αυτή που θα ε, κατακυρώσει το διαγωνισμό να ελέγξει από πού έρχονται τα διάφορα στοιχεία διότι βεβαίως καταρχήν αν πρόκειται για οικοδομή όντως θα έρθουν τα περισσότερα στοιχεία από την αγορά, αλλά αν πρόκειται για ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν ξέρεστε από πού θα έρθουν τα συστατικά τους. Αναρωτιέμαι λοιπόν ότι το άρθρο 6, 6 αυτή η διαδικασία μπορούν να ισχύσουν και μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι εξ αυτές οι αρχές οι οποίες δεν έχουν αρμοδιότητες του ΠΟΕ και δεν μπορούν να ελέγξουν εάν τα προϊόντα όντως παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξουν την εφαρμογή του άρθρου 6 αυτό είναι το βασικό σημείο κατά τη γνώμη μου για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Ε, το άρθρο 8 ε, που είναι το καλύτερο από αυτά που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ε, να εξασφαλίσει, να ενισχυθεί ο μοχλός που θα εξασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους ομολόγους της εάν υπάρχει η πόνη μια μιας απειλής. Αλλά θα ήθελα εδώ να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να δούμε ε, πόσο ε, αναφέρεται αυτή η ε, απειλή στο κείμενο και πόσο θα συνδυαστεί η απειλή αυτή με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ε, πιστεύω ότι η πρόταση ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση αλλά θα, θα απαντήσω και θα σχολιάσω γραπτός το, ε, τη μελέτη των επιπτώσεων και ενδεχομένως ε, φαντάζομαι ότι για τα υπόλοιπα θέματα μπορεί να αναφερθεί και ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Βάιλαρ έχει το λόγο εν ονόματι των ε, ε, σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω στην αρχή μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι στη σελίδα 13 της παρουσίασής της ενδεχομένως ε, είχα αφαιρεθεί, αλλά δεν μπορώ να θυμάμαι ε, αν εδώ αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο κράτος και ευχαρίστως να το ξαναδιαβάσω διότι καλό είναι να έχουμε μία τέτοια, ένα τέτοιο κανονισμό και πρέπει να ξεκινήσω με τα θετικά στοιχεία. Στηρίζουμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα αλλά πρέπει να υπάρχει και εφαρμογή ε, των διεθνών συμβάσεων του ΠΟΕ, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, οι σοσιαλιστές συμφωνούν με όλα αυτά. Πρέπει να δούμε όμως και τη σκοπιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που προσπαθεί να έχει πρόσβαση σε αγορές που είναι τώρα κλειστές και είναι 19% αυτές. Ε, το οποίο ε, ε, νομίζω ότι στο ΑΕΠ τη Ινδίας και άλλων χωρών θα ήταν σημαντικό να μπορέσουμε να εντείνουμε την παρουσία μας. Βέβαια πρέπει να δούμε πώς αυτό θα αναφερθεί σαν υποχρέωση εις την ε, οδηγία διότι λέγεται ότι αν υπάρξουν πολύ χαμηλές προσβολές σε έναν διαγωνισμό είναι είτε επιδοτούμενες τιμές είτε ε, τιμές dumping που αντιμετωπίζουμε από την, από την Κίνα και από άλλες χώρες άρα καλό είναι να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει αν υπάρχουν ε, ε, ε, δυσκολίες προσβάσεως και αν σε ορισμένες χώρες ε, οι δημόσιες προμήθειες όπως παραδείγματος χάρη ε, για το σιδηρόδρομο δεν απελευθερώνονται πράγμα το οποίο επηρεάζει και τις δημόσιες προμήθειες. Το κάνουμε ε, και στην Ευρώπη και είναι νόμιμο για αυτές τις χώρες. Αυτά ήταν τα θετικά. Έχω όμως μια μεγάλη επιφύλαξη και σε αυτήν θα φτάσω τώρα. Διότι στο τελευταίο σημείο του κειμένου σας πιστεύω ότι δεν είναι σωστό και νομίζω ότι δεν το θεωρεί σωστό ούτε η πολιτική μας ομάδα για ε, την αντιμετώπιση της Ευρώπης. Ε, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Ε, δεν πρέπει να λέμε by European αλλά by fair and correct όχι μόνο δηλαδή. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι αν ε, διαφοροποιείται ε, την καναδική και αγορά και την αγορά των ΙΠΑ που είναι πολύ βιομηχανοποιημένες και αν τη συγκρίνεται με την Ινδονησία και ε, την Μιαμάρ που είναι τελείως διαφορετικές διότι ξέρουμε ότι εντωμεταξύ η βιομηχανία είναι πολύ επιφυλακτική για την πρόταση αυτή πάντοτε ενδιαφέρεται για νέες αγορές αλλά αν υπάρξουν αυστηροί περιορισμοί μπορούν να υπάρξουν επιπτώσεις για τις αγορές μας που προσπαθούν να προωθήσουν οι ε, ε, επιτροπή μας και δεν θα υπάρχει η σωστή απήχηση. Επίσης θα ήθελα να ξέρω τι κάνατε με την οδηγία σχετικά με τους διαφόρους τομείς οι οποίοι προωθούσε μια διεθνή αντιμετώπιση και με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ε, και ε, τα GPA διότι ε, είμαστε ανοιχτοί. Είναι σωστό ότι κάτι πρέπει να γίνει Υπάρχουν ορισμένες περιοχές και τοπικές αυτοδιοικήσεις οι οποίες κατηγορούν την Κίνα ότι εξασκεί φοβερό ντάμπινγκ, το βλέπετε στην έκθεση Ταραμπέλα αλλά και στην Πολωνία. Υπάρχουν πολωνικοί παροχοί οι οποίοι έρχονται στη Γερμανική και στην ελληνική αγορά με τόσο χαμηλές τιμές ώστε δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το θέμα λογικά. Είναι ίσως κάτι το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί εδώ θα, γίνει, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με την οδηγία εξυγχρονισμού. Τα υπόλοιπα θέματα μπορείτε να μας τα απαντήσετε ή να μας τα στείλετε γραπτός. Ε, Μάρτιν Λόκρεμπεκ αλλά και αλλά ο κύριος Λόκεγκορτ δεν είναι εδώ. Η κυρία Χέντε Ρούλε τότε εκ μέρου των Πρασίνων τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω ορισμένε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτές θα ξεκινήσω, διότι περιέργως δεν μας είπε καθόλου Επιτροπή τι γίνεται στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται στο Συμβούλιο και πώς την εκτιμά, γιατί σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις υπάρχει μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο και αναρωτιέμαι γιατί πρέπει τόσο να δραστηριοποιούμαστε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα ε, αντικείμενο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο και το Συμβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει αλλά και εγώ έχω και ερωτήματα και προβλήματα γιατί αν διάβασα σωστά την ανάλυση σας ε, είναι μία σαφής προώθηση της εμπορικής πολιτικής ε, και της πολιτικής εξαγωγών, όχι όμως της πολιτικής για τις ε, δημόσιες προμήθειες που είναι ένας νέος όρος τον οποίο δεν ήξερα μέχρι τώρα ε, διότι αυτός ο όρος δεν εφαρμόζεται στην εσωτερική αγορά, ε, εφαρμόζεται στην εξωτερική αγορά και στην την αγορά των εξαγωγών. Οπότε ε, υπάρχουν πολιτικοί στόχοι και σκοπιμότητες που επιβαρύνουν και καθιστούν αυτή την πολιτική πιο δαπανηρή και οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να αναλυφθούν ε, αύριο από τους Ευρωπαίους πολίτες διότι βλέπουμε ότι τώρα οι δημόσιες πωλήσει επιβαρύνονται ε, για το διαγωνισμό με 30.000 ευρώ επιπλέον χωρίς να έχουμε καν την νομική υποδομή ε, πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει περαιτέρω τη διαδικασία. Επίσης όσον αφορά την ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων δεν κοιτάξατε καθόλου το θέμα της ανάθεσης γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος ε, Σβάμπ αν κάποιος αγοράζει ηλεκτρονικούς είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει από πού έρχονται τα διάφορα ανταλλακτικά ή για ε, ε, μηχανές ε, για τα αυτοκίνητα δεν ξέρουμε από πού έρχονται τα ανταλλακτικά είναι μια πολύ περίπλικη και δύσκολη κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε και μου δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την ε, εμπορική πολιτική. Η κυρία Βάιλερ πολύ σωστά είπε ότι στην εμπορική πολιτική πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ ε, των εμπορικών ομολόγων. Αυτό όμως δεν επιτυχάνεται με αυτό το στόχο. Είτε πρόκειται για την Ιαπωνία, είτε για τη ΣΥΠΑ, ή την Κορέα, ή ε, την, τον Καναδά που τίθενται σε ίση βάση με τις υποανάπτυξη χώρες παρόλο που υπάρχει ίσως κατάχρηση ε, των δημοσίων προμηθειών για την εμπορική πολιτική. Κύριε κυρία Μακάρκιν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και με τους ε, συναδέρφους. Μετά πάντως της ε, παρουσίας που ακούσαμε σήμερα, ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά μερικά παραμένουν, μερικές απορίες παραμένουν. Αυτά που ακούσαμε την προηγούμενη φορά από την Επιτροπή δεν φαίνεται να προχώρησαν. Εδώ η ένσταση εξακολουθεί να ισχύει από αυτά που είπατε κι εσείς. Η έκθεση αντικτύπου ήταν πολύ αρνητική. Είπατε ότι η ανάλυση για την ανάγκη και για την αναλογικότητα είναι κάτι που παραμένει ιδιαίτερα αδύναμο και ότι η έκθεση αντικτύπου δεν κατάφερε να πείσει για την αναλογικότητα. Μια τέτοια πολιτική λοιπόν τελικά αφήνει στο διαφερόμενο τη δυνατότητα να επιλέξουν. Θέλω να πω ότι ο κανονισμός τελικά δεν θα ανταποκριθεί στις δικές μας ανάγκες. Δεν καταφέρνουμε να έχουμε ένα πραγματικό μέσο για τις ε, προμήθειες ε, απ' έξω. Τελικά θα είναι αρνητική η γνωμοδότηση γιατί υπάρχουν ε, νομικές αδυναμίες. Οπότε, κατόπιν όλων αυτών, αφού είναι αρνητική η κατάσταση, γιατί η Επιτροπή πιέζει να προχωρήσει. Επειδή κάποιοι το επιθυμούν, ή επειδή πράγματι πιστεύει ότι στην πράξη μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί βλέπετε όλοι θέλουμε να υπάρξει άνοιγμα ε, των ε, αγορών στις τρίτες χώρες και μπορεί να συμφωνεί και το Συμβούλιο με αυτό, αλλά πιστεύω ότι η πρόταση που έχουμε εδώ μπροστά μας σήμερα δεν είναι το σωστό μέσο για να το πετύχουμε. Αν ε, λοιπόν θέλουμε την αμοιβαιότητα, Μήπω τελικά κλείσουμε αντί να ανοίξουμε ευκαιρίες και θα αυξήσουμε τον προστατευτισμό, κάτι το οποίο είναι πολύ αρνητικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν παρουσιάζω τις σοβαρές μου επιφυλάξεις και περιμένω τις απαντήσεις σας. Η κυρία Ρίτοβα ίσως θέλει και εκείνη το λόγο, ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οφείλω να σας πω ότι την ιδέα αυτή εγώ τη βρίσκω απολύτως ορθή. Γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να δημιουργηθεί αμοιβαιότητα. Όχι τόσο για αυτές καθεαυτές τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά γενικότερα για τις ε, ανταλλαγές, τις εμπορικές γιατί υπάρχει η εμπορική μα πολιτική και υπάρχει και ο μηχανισμός αυτό για τις δημόσιε συμβάσει. Άρα είναι αυτό το κατάλληλο μέσο για να πετύχουμε την αμοιβαιότητα. Η γενική ιδέα δηλαδή πιστεύω ότι είναι ορθή, αλλά ο τρόπος που τη χειριζόμαστε πιστεύω ότι δεν είναι σωστός. Αν δούμε την επιλογή 3β, τελικά πώς θα λύνονται σε αυτή την περίπτωση τα προβλήματα από τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την βούληση ή την έλλειψη βούλησης αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι διέπουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις σε έναν βαθμό και δεν καταλήγουν ποτέ σε συμπεράσματα. Δεν καταλήγουν γενικά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο ή τέλο πάντων τι μηχανισμός θα χρειάζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές θα καταλήγουμε σε κάποια απόφαση αντί να κλείνουμε την αγορά μας. Πώς θα πετύχετε όλες οι χώρες μέλη σε περίπτωση που ληφθεί τέτοια απόφαση να κλείνουν πράγματι τις αγορές τους, αν έτσι πρέπει, αν έτσι αποφασιστεί. Θα συνεχιστούν διαπραγματεύσεις για χρόνια ακόμα ή φαντάζεστε να υπάρξει κάποια λύση ή θα δημιουργήσετε ένα διεθνές σώμα για τις μεγάλες ε, οικονομίες του κόσμου στις οποίες θέλουμε να δυσδύσουμε και αυτή η Διεθνής Αρχή θα λειτουργεί σαν ε, διαιτητικό σώμα. Πώς θα ελέγξουμε την πρόσβαση στις αγορές ε, αυτές που είναι πολύ σημαντικές για μας. Αυτό για μένα είναι σημείο κλειδί στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρθηκε ήδη, που έχει να κάνει με τους Δήμους ή τέλο πάντων με τα σώματα, τα όργανα εκείνα, τα οποία δεν έχουν ε, αρκετό διοικητικό προσωπικό. Οπότε πώς ε, θα καλυφθούν περιπτώσεις υπερεργολαβίας ή πώς θα εξηγήσετε ότι ακόμα και για τα αγαθά που δεν καλύπτονται θα χρησιμοποιούνται κάποια κανάλια μέσω ενός Ευρωπαίου ε, Ευρωπαϊκής Αναθέτουσας Αρχής που θα χρησιμοποιεί κάποιον υπεργολαβικά. Αυτά προς το παρόν. Φυσικά παραμένουν και άλλα ερωτήματα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αν καταφέρουμε να φτάσουμε σε λύση, αυτό θα είναι μάλλον ένας κανονισμός παρά μια οδηγία για μένα. Ευχαριστούμε κυρία Ρωτήκο. Βάλλος κανείς από τους ευρωβουλευτές θέλει το λόγο. Όχι. Οπότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω και θα ζητήσω από τον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς να απαντήσει. Πιο πολλοί σχόλια ακούσαμε παρά ερωτήσεις. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε και θα απαντήσουμε ατομικά στους ευρωβουλευτές για κάποια από αυτά τα ζητήματα αν δεν καταφέρω τώρα να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ό,τι συζητήσεις και αν έγιναν μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε τις διαδικασίες στο εσωτερικό της Επιτροπής που έγιναν να σας τις αναφέρουμε λεπτομερώς. Είναι θέμα του συλλογικού σώματος της ε, Επιτροπής. Έτσι δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για την ε, έκθεση αντικτύπου. Πολύ σύντομα. Έγιναν δύο έτσι καλώς είναι το περισσότερο που μπορεί να προβλεφθεί. Άλλαξαν πολλά πράγματα προκειμένου να ληφθούν ε, υπόψη λοιπόν τα συμπεράσματα της έκθεσης αντικτύπου. Και τελικά το σώμα των επιτρόπων ανέλαβε την ευθύνη και αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση ως είχε. Και δεν υπάρχει νομική γνωμοδότηση νομικά εμπόδια. Τώρα είναι και το Συμβούλιο που θα το δει. Τώρα κάποιο ρώτησε ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο. Δεν σα κρύβω ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο είναι δύσκολη επί του παρόντο. Υπάρχει μια διαφωνία, περισσότερη είναι κατά, αλλά μόνο δύο συζητήσεις έγιναν προκαταρτικά στην ομάδα εργασίας. Οπότε είμαστε πολύ νωρίς ακόμα για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τις προπτικές που έχει η πρόταση αυτή να περάσει στο Συμβούλιο δεν εξετάστηκε καν εξ η πρόταση ακόμα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση όταν, αν μη τι άλλο, θα έχουν συζητηθεί όλα τα θέματα στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Στην πράξη τώρα, πώς θα προχωρήσει αυτό. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και βάζουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα βήματα, για την κεντρική διαδικασία έτσι κι αλλιώς έχει πάρει κοινοποίηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μείνει σε κρεμότητα επάπειρο. Τα άρθρα 8 και 10 αποτελούν μέρος της πρότασης και η ιδέα είναι πάντα να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερες πιθανότητες να λυθούν στις διαπραγματεύσει τα προβλήματα. Γι' αυτό και αφήνουμε αρκετό χρόνο. Η Επιτροπή χρειάστηκε 9 μήνες για να ερευνήσει και είναι νομίζω 12, όσο πέντε μήνες για τις διαπραγματεύσει προβλέπονται. Υπάρχει λοιπόν χρονοδιάγραμμα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σέρνεται το θέμα πάπυρο. και αυτό το μήνυμα στέλνουμε. Και έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει εφόσον χρειαστεί. Για τις συγκεκριμένες τώρα διαδικασίες καθορίζονται ξεκάθαρα τι ισχύει για την ε, πλειοψηφία που μπλοκάρει την απόφαση. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε ε, λύση μετά από διαπραγματεύσεις. Οι προτάσεις σας είπα μόλις έχουν φτάσει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο παίρνουμε κάποια μηνύματα από τρίτες χώρες ότι η Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, μας θύμισαν, έχει, σκέφτεται το θέμα της, ε, του να είναι μέλος ή όχι. Θα υπάρξουν δηλαδή επιρροές και εκτός σε άλλες χώρες. Οι χώρες θα επηρεάσουν την εξέλιξη της διαδικασίας. Ήδη από τώρα. Έτσι κι αλλιώς εμείς πάντα λέμε στα τρίτα μέρη να κάνουν κάποια βήματα για να ανοίξουν την αγορά τους ήδη από πριν. Υπάρχει διάκριση τώρα σε χώρες όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, αναπτυγμένες οικονομίες δηλαδή, η Ιαπωνία και ο Καναδάς. Η πρόταση αποκλείει τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Εκεί δεν ε, μπορεί να υπάρξει μέτρο διάκρισης, δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο μέτρο δηλαδή για αυτές τις χώρες. Έτσι κι αλλιώς ε, διαβαθμισμένη θα είναι η προσέγγισή μας. η κατάσταση είναι διαφορετική αν μιλάτε για μια οικονομία σαν εκείνη της Κίνας ή για άλλες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Πάντα για τον αντίκτυπο και για αυτά που γνωρίζουμε όσον αφορά τις εμπορικέ συμφωνίες, FTAs. Το πρόβλημα που βλέπουμε είναι ότι από την άλλη μεριά του τραπεζιού ακούμε ότι πιστεύουν πως την πρόσφασή τους πρέπει να την παίρνουμε σε κάτι το δεδομένο. Δηλαδή θεωρούν ότι ήδη το δικαιούνται. Αυτό είναι που δημιουργεί προβλήματα στις διαπραγματεύσεις, γιατί αρχίζουν να ε, βλέπουν ε, τη διαπραγμάτευση σε άλλα σημεία και όχι εκεί, γιατί αυτό το θεωρούν και εκτιμένο ήδη. Προσπαθούν να κερδίσουν δηλαδή σε άλλα σημεία στη διαπραγμάτευση αντισταθμίσματα δηλαδή αλλού. Εμείς δεν βλέπουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει σε μια κατάσταση όπου δυναμικά να πρέπει να πληρώσει δύο φορές για το άνοιγμα αυτό της αγοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Δεν μπορεί η άλλη πλευρά να θεωρεί δεδομένο κάτι το οποίο για μας είναι στη διαπραγμάτευση και το διαπραγματευόμαστε. Αλλιώ γίνονται πάρα πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Για το άρθρο 6 ακόμα υπάρχει κάτι, για να δω τι άλλο έχω εδώ. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Έτσι κι αλλιώς αν κάποιος θέλει επιπλέον εξηγήσεις ή αισθάνεται κάποιος ότι δεν απάντησα στην ερώτησή του, παρακαλώ, συνάδελφος τώρα. Για το άρθρο 6. Η ερώτηση ήταν, ε, οι αρχές, πώς θα ξέρουν πότε πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς. Μα πρέπει να εφαρμόζουμε τον τολωνιακό κώδικα έτσι κι αλλιώς. Τώρα ρωτάτε πώς θα εφαρμόζουμε αυτό το κώδικα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εδώ πέρα ότι μιλάμε και για την, το τελευταίο στάδιο μεταποίησης για να ξέρουμε από πού έρχεται το αγαθό. Αν πρόκειται για κομμάτια, για κομπιούτερ, τα οποία έρχονται από άλλες χώρες αλλά συναρμολογούνται, στην Ευρώπη, τότε θεωρείται ευρωπαϊκό αγαθό. Αφού προηγουμένω δούμε πόσα είναι τα κομμάτια τα οποία αποτελούν αυτό το ανταλλακτικό. Έπειτα, για το άρθρο 6 πάντα. Είναι προαιρετικό μέσο. Οι αρχές που δεν θέλουν να εμπλεκτούν σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι υποχρεωμένες. Οι τρίτες πλευρές επίσης όταν αρχίζει η διαδικασία υπάρχει μια δήλωση από τους προμηθευτές με διευκρίνηση. Ακόμα και αν μια αρχή πει ότι θέλει να μπλοκάρει, εμείς πρέπει να το ελέγξουμε αυτό στη συνέχεια. Για την ερώτηση της κυρίας Βάλ για το ποιες χώρες μέλη δεν είναι κυκλισμένον των ε, θυρών η σε αυτή και γι' αυτό και δεν αναφέρθηκα σε χώρες μεμονωμένα. Άμα θέλετε γραπτά μπορώ να σας δώσω την απάντηση που ζητήσατε. Πρόεδρος, ευχαριστώ και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Έτσι έληξε η συνεδρίασή μας. 11 και 12 Οκτωβρίου θα τα ξαναπούμε.